και οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις τρίτες χώρες οι οποίες εμπλέκονται. Και πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο δράσης τονίζει ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ικανότητος, γιατί η έλλειψη ικανότητας εφαρμογής εμποδίζει την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας μεταναστών και την ίδια τη συνεργασία. Και κάνουν αδύνατο να υπάρξει δίωξη των ε, διακινητών σε όλη την αλυσίδα διακίνησης των μεταναστών. Με το σχέδιο λοιπόν δράσης, η Κομισιόν έχει σαν στόχο να δώσει τεχνική και οικονομική βοήθεια στις τρίτες αυτές χώρες, ώστε να υποστηριχτεί η ανάπτυξη εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για να αντιμετωπιστεί η λαθρεμπορία μεταναστών και να δημιουργήσουν πολιτικές κατά της διαφθοράς που οδηγούν σε προβλήματα για την διακίνηση μεταναστών και να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης το οποίο θα μειώσει το φαινόμενο αυτό. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την Τουρκία έχουν, πρωτα... έχουν αναλυφθεί ήδη ορισμένε διαρθρωμένε δράσεις στο παρελθόν για να υποστηριχθεί η προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τις απαραίτητε ικανότητε σε θέματα εσωτερικών. Έχει δοθεί χρηματοδότηση επί τη βάση του προενταξιακού εργαλείου στον τομέα των εσωτερικών και θα δοθούν περισσότερες ε, αρρωγές τα επόμενα χρόνια. Επομένως, με όλα αυτά είναι φανερό ότι η Κομισιόν συμμερίζεται τις ανησυχίες του μέρους του Κοινοβουλίου σε σχέση με την ανάγκη να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες για να αντιμετωπίσουμε τη λαθρεμπορία μεταναστών και συγκεκριμένα με την Τουρκία. Η γραπτή απάντηση στο κοινοβουλευτικό αυτό ερώτημα θα, θα διατυπωθεί πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα κάνουμε συζήτηση. Έχουμε λάβει την απάντηση της εκπροσώπησης της Κομισιόν. Θα περάσουμε όμως όπως ελέγχθη προηγουμένως αιτήσει της ομάδας των Πρασίνων σε μια συζήτηση για την <clears throat> κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία. Όπως ξέρετε 1η Νοεμβρίου θα λάβουν χώρα εκλογές σε ένα κλίμα όλο και πιο ακραίας πόλωση σε πολιτικό επίπεδο. Είχαμε το τη δρομοκρατική επίθεση στο Σιουρίκ που οδήγησε στο θάνατο 34 ε, ανθρώπων από ένα μέλος του Ισλαμικού κράτους, αλλά έχουμε και τις ενέργειες του ΠΚΚ, τις βίες αυτές ενέργειες. Η βία είναι πολύ δύσκολη και πολύ έντονη στα νοτιοανατολική Τουρκία, διότι δηλαδή στα σύνορα της Συρίας με δεκάδες θυμάτων. Η τουρκική κυβέρνηση έχει κηρύξει στρατιωτική ζώνη την περιοχή αυτή και έχει αναστείλει ορισμένες ε, ε, ελευθερίες και έχουν υπάρξει επιθέσεις κατά του Χαντεπέ και των γραφείων της εφημερίδας Χουριέτ. Θα δώσουμε το λόγο στον Χαβιέ Νίνιο Πέρες, ο οποίος είναι ο υπεύθυνο της ε, εξωτερικής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για την Τουρκία και μετά για τον αρμόδιο για τη διάμεση. Καταρχήν ο κύριος Χαβιέ Νίνιο Πέρες. Συγγνώμη, συγγνώμη. Θα απαντήσουν μετά τη συζήτηση, δεν θα λάβουν τον λόγο εξ αρχής. Οπότε μπορείτε να θέσετε ερωτήματα και να σχολιαστεί. Κύριε Πύρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους πρασίνους που προσέθεσαν το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Ε, μέσω του αιτήματό Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι όπως είπε και ο Πρόεδρος βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ένας φαύλος κύκλος βίας ε, όπου κανείς πλέον δεν έχει τον έλεγχο. Απ' τη μια βλέπουμε τις επιθέσεις του ΠΚΚ μέσα σε μια εβδομάδα κατά 14 ε, ε, αστυνομικών, 16 στρατιωτικοί πέθαναν και βλέπουμε και φυσικά και τα αντίπεινα από την κυβέρνηση με την κατάσταση στο Τσίστρε που ήταν πολύ κρίσιμη για 19 ημέρες. Η κουρδική αυτή πόλη ήταν ε, ε, μπλοκαρισμένη τελείως, ε, υπήρχε ένα καθεστώς επιτήρησης και φοβάμαι πολύ ότι διότι η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ κρίσιμη και ευαίσθητη. Και είδαμε και στην Ευρώπη και στις πόλεις μας διαδηλώσεις εχθές και στο Ρότερνταμ και στο Άμστερνταμ είχαμε μεγάλες διαδηλώσεις και είδαμε και εντάσεις μεταξύ ε, Κούρδων και Τούρκων και στα κράτη μας και στις κάτω χώρες και στο Βέλγιο και επομένω όταν υπήρξε η έκκληση αυτή από τις πολιτικές ηγέτες όλων των πολιτικών κομμάτων να ζητούν να περιοριστεί η βία ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάπου να σταματήσει όλη αυτή η βία. Βλέπουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών ε, κομμάτων, ε, κυρίως του ΧΑΝΤΕΠΕ που ε, υπήρξε αντικείμενο επιθέσεων 304 άνθρωποι μέλη του ΧΑΝΤΕΠΕ υπήρξαν αντικείμενο επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα και δυστυχώς το τελευταίο εξάμεινο διαπιστώνουμε ότι όλα όσα είχαν επιτευχθεί μέχρι τούδε πλέον έχουν απομακρυνθεί εντελώς και έχουν ανατραπεί. Ε, επιθέσεις ε, κατά μέσω μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο κατά της ε, Χουριέτ, αλλά και κατά της ημερησίας Σαμπά, ξένοι δημοσιογράφοι στις κουρδικές περιοχές δεν έχουν καμία δυνατότητα να κάνουν μεταδόσεις και να γράψουν για το τι συμβαίνει και υπάρχει θέμα ελευθερίας του τύπου. Πρέπει λοιπόν και εν ώψη των εκλογών να ρυθμιστεί το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου. Ε, ένα τελευταίο για τη μετανάστευση, διότι συζητήθηκε ήδη και πρόκειται για ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους όταν συζητούμε για την Τουρκία. Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται κατά νου είναι η μετανάστευση. Ποιοι είμαστε εμείς βέβαια οι οποίοι ε, θα κατηγορήσουμε την Τουρκία που τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει υποδεχθεί δύο εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν λόγοι να συζητούμε. Να συζητούμε για το η λαθρεμπορία, για παράδειγμα, την οποία συζητήσαμε προηγουμένω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το θέμα είναι πώ μπορούμε να βοηθήσουμε και την Τουρκία περισσότερο, προκειμένου να υπάρχει αυτά τα δύο εκατομμύρια προσφύγων που βρίσκονται επί τόπου. Δεν είναι μόνο το θέμα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και το πώς μπορεί να βοηθήσει η Τουρκία εμάς, αλλά και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε την Τουρκία. Και πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και ιδέες και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν να μην υπήρξε έκκληση σε πολιτικό επίπεδο σε υψηλό πολιτικό επίπεδο για διάλογο με την Τουρκία για το θέμα της μετανάστευσης. Επίγει το ζήτημα. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, ίσως ε, για μας ως Επιτροπή Εξωτερικών Επιθέσεων. Με αυτό το, το φαύλο κύκλο βία που έχει ξεκινήσει τώρα στην Τουρκία. Θα ήθελα εμεί ω Επιτροπή να καλέσουμε, παρά το γεγονό ότι πρόκειται για υπηρεσιακή κυβέρνηση, ε, τον ε, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων τη Τουρκία να έρθει εδώ για να μιλήσουμε για το τι ακριβώ συμβαίνει στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Και όντως είναι πολύ καλή αυτή η ιδέα και θα ήθελα να το πω και εγώ αυτό. Ο κύριος Τζαμπάσκη έχει το λόγο. It sounds like Τζαμπάσκη. Ωραία. <laughs> Уважаеми колеги, уважаеми представители на... Αγαπητοί συνάδελφοι, Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τουρκική κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή περίπου 20% του πληθυσμού της Τουρκίας. Ξέρουμε ότι οι κουρδικές θέσεις στο βόρειο Ιράκ και στη βόρεια Συρία υφίστανται επιθέσεις και η Τουρκία με τον τρόπο αυτό έμεσα βοηθάει το Ισλαμικό κράτος. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια συνενοχή κάποια συμπερνία μεταξύ Τουρκίας και Ισλαμικού κράτους. Έχει φτάσει η Τουρκία να πολεμάει τους δικούς της πολίτες για να εμποδίσει τους Κούρδους να έχουν μια καλύτερη στατική θέση γιατί επίκεινται οι εκλογές και ο Ερντογάν θέλει να πάρει την πλειοψηφία των ε, ψήφων. Εγώ ως Βούλγαρος βλέπω ότι η Τουρκία οργανώνει την διακίνηση μεταναστών που έρχονται σε εμά. Όλοι αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν από κοντά τα θέματα αυτά το γνωρίζουν. Γι' αυτό θα ήθελα να έχω μια σαφέστερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. <clears throat> Ίσως πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και όχι να προσπαθούμε να εθελοτυφλούμε σε ένα πρόβλημα που είναι πραγματικά τραγικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Η κυρία Ζώμερα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σκεφτούμε και λίγο περισσότερο για το ρόλο του Πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα έχει μονάχα ένα επίσημο ρόλο, αλλά από ό,τι βλέπουμε από τα νέα, από τις ειδήσει, έχει φτάσει να παίζει ένα πολιτικό ρόλο να απειλεί όχι μόνο το ΠΚΚ αλλά και όλους τους Κούρδους και να απειλεί το ΧΑΝΤΕΠΕ το οποίο πια δεν θα είναι σε θέση ουσιαστικά να κάνει προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές λόγω της κατάστασης στην Νοτιοανατολική Τουρκία. Έχει κάνει στην εντύπωση ότι στην Τουρκία έχει εξαπολυθεί μία μορφή βίας που περιλαμβάνει και την υποστήριξη της κυβέρνησης για να στρίψει, να στρέψει μάλλον τις εκλογικές προτιμήσεις των πολιτών προς την κατεύθυνση που επιθυμεί η κυβέρνηση. Εγώ βρίσκω πολύ θετική την ιδέα να προσκαλέσουμε τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων της ε, Τουρκίας και να μπορέσουμε να του θέσουμε ερωτήματα. Μπορούμε και τον ε, πρεσβευτή να καλέσουμε να θα μας πει τα ίδια και τα ίδια. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το τεράστιο κύμα προσφύγων που έρχονται προς την Ευρώπη και το ερώτημά μου είναι πώς έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μας. Η δική μου εντύπωση είναι ότι έρχονται όλοι από, πολλοί από αυτούς από την Τουρκία και τι γίνεται τώρα με την συμφωνία επανεισδοχής που έχουμε ε, υπογράψει. Επίσης υπάρχει η φήμη ότι η Τουρκία στέλνει η ίδια τους πρόσφυγες προς την Ευρώπη. Έχει στα σύνορά της προς την Συρία δύο εκατομμύρια πρόσφυγες και γι' αυτό από εκεί προέρχεται η μεγάλη μάζα των προσφύγων προς την Ευρώπη. Θα ήθελα εδώ να έχω λοιπόν την ε, άποψη του εκπροσώπου της ε, τουρκικής κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Προφανώς πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και έχουμε και υποχρέωση ως ε, Ευρώπη να βοηθήσουμε την Τουρκία. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο οργανωμένο και όχι άναρχο. Κύριος Χατζηγεωργίου. Ε, έχουν δίκιο οι συνάδελφοι που έχουν πει ότι χωρί την παρουσία ενό εκπροσώπου τη τουρκική κυβέρνηση εδώ, εγώ θα πρότεινα τον Υπουργό Εξωτερικών. Ουσιαστικά η συζήτηση μα έχει βέβαια αξία, αλλά μειωμένη σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να μάθουμε ή να πούμε ε, στην παρουσία είναι Τούρκου αξιωματούχου. Η, Τουρκία, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι φανερό ότι είναι στα όρια του χαου Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προέβλεψε τι εξελίξεις όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στη γύρω περιοχή. Δεν πρόβλεψε ότι οι πόλεμοι θα έφερναν όλο αυτό το τσουνάμι του προσφυγικού κύματο και σήμερα πολλές χώρες που ουσιαστικά ενεπλάκηκαν σε αυτή την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, να σας θυμίσω ότι έτσι τη χαρακτηρίζαμε όλοι εδώ, πολύ λίγοι από εμά έλεγαν ότι έρχεται Αραβικός χειμώνας, γιατί βλέπαμε και αναλύαμε καλύτερα το τι έτρεχε στις χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας. Ε, σήμερα, εν πάση έχει ουσιαστικά καταρακωθεί η προσπάθεια επίλυσης του κουρδικού προβλήματος. Ε, εγώ σαν Ευρωβουλευτής από την Κύπρο έχω, αντιλαμβάνεστε, αυξημένη ανησυχία για το τι τρέχει στην Τουρκία, γιατί μας επηρεάζει άμεσα, αλλά και η καταστροφική εξέλιξη στην επίλυση του κουρδικού επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να απασχολεί όλους. Ε, θέλω να σας πω ακόμα ότι πολλοί αναλυτές λένε ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος Ερτογάν αν δεν δημιούργησε, επέτρεψε ε, τις ε, εξελίξεις αυτές, ακόμα και τις συγκρούσεις και τις δολοφονίες, τις άφησε να συμβούν δηλαδή, κρίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η ανασφάλεια των πολιτών και αυξανωμένη της ανασφάλειας των πολιτών θα επανακάμψουν στο, στο κόμμα του στις επικείμενες εκλογές της πρόεδρου του ε, επίσης αυξάνοντας το εθνικό εγώ, όταν ένα κράτος βρίσκεται σε τέτοια αναταραχή αυξάνεται το εθνικό εγώ, όπως το λέω, και πάλι αυτό σπρώχνει προς την, ε, να αυξηθούν οι ψήφοι του κυβερνώντος κόμματος, σε μια εντύπωση σταθερότητας. Ε, αντιλαμβάνεστε τώρα όταν στην αρχηγία ενός κράτους βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος ε, συμπεριφέρεται κατά πολλούς αναλυτές και κατά τη δική μου άποψη με έναν τρόπο τέτοιο ανεξάρτητα από το το αίμα που τρέχει, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξημένο, πολύ πολύ αυξημένο ρόλο να διαδραματίσει, έστω και σχετικά αργά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ και θα ήθελα ξεκινώντας να αναφερθώ σε αυτά που είπε και η Κάτι Πύρη και να ευχαριστώ και την κυρία Ζόμερ. Θα ήταν καλό να προσκαλέσουμε τον Υπουργό των Εξωτερικών και είναι της υπηρεσιακής κυβέρνησης στην Επιτροπή μας και καθώς έχω προτείνει και εκ μέρους του Πρασίνου να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια θα έλεγα μια συζήτηση ε, μαζί του να ακολουθηθεί και από συζήτηση στην Ολομέλεια γιατί η κατάσταση δεν θα αλλάξει γρήγορα. ήταν απαραίτητο. Έρχονται και οι εκλογέ. Επίση, συμφωνώ με εκείνου που λένε ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση όχι μόνο για τη μετανάστευση. Θα πρέπει να γίνει σύνοδο κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Η κατάσταση αναφέρθηκε ο Ερντοάν νωρίτερα, στην οποία βρίσκεται και τα όσα κάνει τα τελευταία χρόνια, καταστρέφει αυτά για τα οποία αγωνιστήκαμε όλοι εμείς που δεν έχουμε σχέση με ε, θρησκευτικές οργανώσεις. Άνοιγμα. Η κατάργηση της κατάστασης εκτακτής ανάγκης είναι τελείως αντίθετα από αυτά τα πράγματα αυτά που κάνει τώρα. Και δεν αναφέρομαι και στις επιθέσεις κατά των Κούρδων και όχι μόνο του ΠΚΚ, κατά γραφείων του HTP, 304 λέει τις τελευταίες εβδομάδες, εις βάρος πολιτών Κούρδων στο Ντίτζρε, με πολλούς νεκρούς αμάχους, απαράδεκτο. η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι μας, όλοι όσοι έχουμε αυτές τις θέσεις και στο Συμβούλιο, πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι ο Ερντοάν και η Τουρκία αποδίονται σε πόλεμο στο πλευρό μας κατά του Ισλαμικού κράτους. Δεν κάνει αυτό ο Ερντοάν και δεν κάνει αυτό η Τουρκία. Ο Ερντοάν αποδίεται σε πόλεμο κατά του ΠΚΚ με την, όπως την νοεί ο ίδιος ε, έννοια του εχθρού μέσα στο τουρκικό κράτος. Και δεν είναι τρόπος αυτός για να καταπολεμήσει το ΙΕΣ, ούτως ή άλλως το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Απέχει πολύ και για τη μετανάστευση. Συμφωνώ με όλους εκείνους που λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να υποστηρίξουμε ε, τους καταβλισμούς των προσφύγων και την κατάσταση που αντιμετωπίσουν όχι μόνο στην Τουρκία βέβαια αλλά και στην Ιορδανία και τον Λίβανο όπου εκατομμύρια προσφύγες έχουν ήδη βρει καταφύγιο ε, από την ύπατη από το πρόγραμμα για τα τρόφιμα, ό,τι και να γίνεται δεν είναι σωστός τρόπος να δοθεί βοήθεια. Πρέπει να βρούμε λύσεις στους πρόσφυγες επιτόπου. Και επίσης, όπω είπε ο κύριος Βαλέρο νωρίτερα σε άλλη συζήτηση, το να θεωρείται ασφαλής χώρα προελεύσεως για πρόσφυγες η Τουρκία, δεδομένη της κατάστασης που έχουμε τώρα και τον πόλεμο ή εν πάση περιπτώσει μεταξύ των τουρκικών αρχών και κατά των Κούρδων ΠΚΚ κουρδικών θεσμών, HTTP δηλαδή, το κόμμα HTTP, είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά πια, γιατί δεν είναι πια ασφαλής χώρα η Τουρκία ως χώρα προέλευσης. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Λούνατσεκ. Και εγώ είχα ζητήσει το λόγο από τον εαυτό μου, αλλά θα είμαι πάρα πολύ σύντομο και θα υποστηρίξω απλώς αυτά που είπαν οι συνάδελφοι για το τι χρειάζεται. να έρθει ο αρμόδιος υπουργό να έχουμε μια διασύρτηση κορυφής πριν να μιλήσουμε για μια χώρα του ΝΑΤΟ που κατά την άποψή μου έχει παίξει ένα αρνητικό ρόλο όχι μόνο για το Ισλαμικό κράτος αλλά και για την κρίση των προσφύγων. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι αξιόπιστα και τα οποία μιλούν για λαθρεμπόριο που γίνεται από τις ε, τουρκικές αρχές για πετρέλαιο το οποίο παράγεται στις περιοχές του Ισλαμικού κράτους. Και η συμμαχία των, ε, κατά του Ισλαμικού κράτους τελικά φαίνεται ότι στρέφεται τελικά κατά των Κούρδων 1% βομβαρδίζουν το Ισλαμικό κράτος 99% ε, τα 100 που αγωνίζονται εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Γιατί χωρίς, έτσι χωρίς σε δυνάμει δεν μπορεί να κάνει κανεί τίποτα. Δεν μπορεί κανεί να κάνει τίποτα με ένα αερισμό να επιδρομές. Δίνω το λόγο στον κύριο Νίνιο Πρέτο από την Υπηρεσία εξωτερική δράση για πέντε λεφτά. Τώρα για να απαντήσει. Δεν θα χρειαστώ πέντε λεφτά. Να παρουσιάσω τον εαυτό μου, Χαβερνίνιο, από, την, ε, από το τμήμα για την Τουρκία εδώ και μία εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Βλέπω να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χώρα αυτή και προσβλέπω σε μια καλύτερη συνεργασία μαζί σας. Θα παραμείνω λοιπόν στην διάθεσή σας για αυτή τη συζήτηση και σήμερα και στο μέλλον. Τρία κύρια στοιχεία αναφερθήκανε. Πρώτα το θέμα της ασφάλειας και τα πρόσφατα γεγονότα στην Νοτιοανατολική Τουρκία. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω πολλά περισσότερα ή να πω τα πράγματα περισσότερο από αυτά που σας είπε ο πρεσβευτής Χάμπα προηγουμένως ανησυχούμε για την κατάσταση στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα της Τουρκίας να προστατευτεί έναντι των επιθέσεων τρομοκρατικής οργάνωσης, αλλά όπως είπατε πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να είναι αναλογική η απάντηση και θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η αναλογικότητα. Αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ένα κλίμα σταθερότητος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας σε όλη τη χώρα, αλλά φυσικά ιδιαίτερα στην νοτιοανατολική Τουρκία. Δεν νομίζω όμως κάτι άλλο μπορώ να προσθέσω πολλά περισσότερα σε αυτά που είπε ο, ο πρέσβης Χάμπερ. Ένα δεύτερο θέμα που αναφέρει από τους ομιλητές είναι το θέμα της μετανάστευσης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα είναι μόνιμο στην, στο θεματολόγιο, όχι μόνο σε σχέση με την Τουρκία, αλλά και για όλη την περιοχή. Όπως έλεγα. θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για το πώς να βοηθήσουμε την Τουρκία και ο συναδελφός μου από την Γενική Διεύθυνση για τις, ε, την DGNIR από, για τις γειτονικέ χώρες ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με αυτή τη Γενική Διεύθυνση και θα μας πει λίγο, λίγα περισσότερα για το τι μπορούμε να κάνουμε. Και φυσικά το ερώτημα παραμένει για το τι μπορούμε να κάνουμε εν ώψη των εκλογών, τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία και να συνδέσουμε όλα αυτά με την ε, επίτευξη της ασφάλειας. Ο κ. Πατρίκ θα πει λίγο περισσότερο για τα θέματα συνεργασίας, για τα πολιτικά θέματα. Φυσικά όλη η ιεραρχία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης μέχρι και η κυρία Φογκερίνη τα έχουν αυτά στο μυαλό τους. Τρίτο στοιχείο, πώς θα έχουμε μια πιο διαρθρωμένη προσέγγιση με την Τουρκία. Πώς θα αναπτύξουμε καλύτερα τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαδικασία προσχώρησης για μας είναι το καλύτερο εργαλείο για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα. Προσπαθούμε να διευρύνουμε αυτό το πλαίσιο και να έχουμε και επαφές για άλλα θέματα. Αναφέρθηκε στο εμπόριο, την ενέργεια, την ασφάλεια ο κ. Χάμπερ και μιλώντας πολύ ειλικρινά υπάρχουν τομείς όπου συμφωνούμε με την Τουρκία και αλλού που διαφωνούμε. Ως εταίροι όμως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί για τι απόψει μα. Υπάρχει σαφές ενδιαφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με την Τουρκία. Ακούσατε για την πρόσφατη αυτή επίσκεψη και τι άλλες επισκέψει υψηλού επίπεδου. Έχουν γίνει σημαντικέ και ενδιαφέρουσες προτάσεις για να έλθουν οι αρμόδιοι υπουργοί της Τουρκίας στις Βρυξέλλες να υπάρξει μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου θα μεταφέρουμε αυτές τις ιδέες στις, στους αρμόδιους υπευθύνους της Κομισιόν και θα επανέλθουμε με προτάσεις για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νίνιο Πέρες. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Πάτρικ Πάκερ, ο οποίος είναι επικεφαλής του Τμήματος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι εμείς είμαστε εδώ η Αγία Τριάδα, είναι μαζί μας και η Γενική Διεύθυνση HOME για να συζητήσουμε τα διάφορα θέματα για την Τουρκία, για τα οποία συνεργαζόμαστε τους τελευταίους μήνες. Δεν ξεκίνησαν αυτά το περασμένο καλοκαίρι. Ε, υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας όταν ξεκίνησε ο διάλογος για τις θεωρήσεις διαβατηρίων ε, και πέραν αυτού υπήρξε και μια πολύ σημαντική διάσταση της δουλειάς μας ε, για την ε, βοήθεια τα τελευταία 6 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολλά από τα πράγματα της συνεργασίας μας ήδη υλοποιούνται για να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση. Συμφωνώ βέβαια μαζί σας ότι πρέπει να αλλάξει η διάσταση της συνεργασίας μας με την Τουρκία στα θέματα αυτά. Και η ευρωπαϊκή πλευρά άρχισε ήδη να τα συνειδητοποιεί αυτά από την περασμένη άναξη όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρθηκε στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία με την Τουρκία λόγω της κατάστασης στη Συρία και στο Ιράκ κυρίως και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, εμπορίας μεταναστών. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η Τουρκία πρέπει να θεωρείται ως εταίρος και όχι μόνο ως πηγή του προβλήματος, είναι και τμήμα της λύσης. Θα ε, ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η Τουρκία έχει αναλάβει το μεγαλύτερο όγκο της μεταναστευτικής κρίσης στην περιοχή εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι η χώρα ε, που έχει υποδεχτεί τους περισσότερους μετανάστες και πρόσφυγες και είναι και αυτή που έχει τους περισσότερους Σύρους που έχουν ε, ε, φύγει από τη Συρία. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε κατά αυτό και θα πρέπει να το εξετάσουμε και με κάποια ταπεινοφροσύνη και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτά που κάνει η Τουρκία. Τρίτον, ε, δεν αδρανεί όσον αφορά τα νέα φαινόμενα και τις νέες τάσεις στη μετανάστευση. Για παράδειγμα, πέρσι συνεργαστήκαμε με την Τουρκία για να ε, δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το φαινόμενο των ε, σκαφών φάντασμα που χρησιμοποιούνταν, ε, εμπορε, εμπορικά σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνταν για την λαθρέα διακίνηση των μεταναστών και αυτό πλέον σταμάτησε χάρη στη συνεργασία με την Τουρκία. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν μικρά σκάφη τα οποία πλέον ε, διανύουν ένα μικρό, ε, μια μικρή απόσταση και αυτό φυσικά είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε και ακόμα διαπιστώνουμε ότι η ορκική εκτοφυλακή τους τελευταίους μήνες βοήθησε να διασωθούν ε, χιλιάδες άνθρωποι στη θάλασσα. Αυτό λοιπόν δεν είναι ασήμαντο, είναι τεράστιο το ποσό. 134 άτομα μόλις διασώθηκαν εχθές. Δεν θα πρέπει λοιπόν να κοφεύουμε και να μην είμαστε εμεί διατεθειμένοι να αλλάξουμε στάση. Ε, ακόμα και το γεγονός ότι οι τουρκικές αρχές ε, πλέον ε, έχουν ε, πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν λόγω της κατάστασης γιατί δεν επαρκεί το προσωπικό τους και επομένως θα πρέπει να δούμε και εμείς να, ε, πώς μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερη βοήθεια και πώς μπορούμε να κλιμακώσουμε τη βοήθεια για την υποδοχή των προσφύγων και προσπαθούμε να συνεργαστούμε ε, από όλους τους πιθανούς διάβλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται λοιπόν το σημείο αυτό, παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι θα ξανασυζητηθεί λόγω της ευαρότητας των όσων συμβαίνουν στην περιοχή και να περάσουμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων για τις τοπικές εκλογές στην Αλβανία, τοπικές εκλογές οι οποίες έγιναν στις 21 Ιουνίου και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 29 έκτου συμφώνησε να προσκαλέσει την επικεφαλή της αποστολής ε, των εκλογικών παρατολιτών και την πρέσβυρα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία. Καλωσορίσω λοιπόν ε, την κυρία Όντρι Κλόβερ που είναι επικεφαλής της αποστολής ε, των εκλογικών παρατηρητών του ΑΣΕ και την πρέσβυρα Ρωμάνα ε, Βλαχούτιν που είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία και να καλωσορίσω και την κυρία Μπαέατα Μαρτίν Λόβικ που είναι επικεφαλής του τμήματος εκλογικών του ΑΣΕ ε, γάμα δέλτα θήτα δέλτα. Έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα της παρατήρησης. Ε, θεωρείται ότι οι εκλογές έγιναν ε, με κατάλληλο τρόπο. Η προεκλογική εκστρατεία ήταν ήρεμη και η τελική έκθεση επιβεβαιώνει μία σειρά αποθετικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη ε, υπήρξαν συγκεκριμένε ε, διαδικασίες οι οποίες στηρίθηκαν, ε, κάποιες αμφισημίες, κάποια νομικά ε, ζητήματα, κάποιες καταγγελίες εξαγοράς ψήφων και υπήρχαν και κάποιες ε, καταγγελίες που ίσως παρακολύουν τις τη διεξαγωγή των πραγματικών εκλογών. Αυτό θα έπρεπε να το απασχολήσει φυσικά τις αλβανικές αρχές, αλλά θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τις κυρίες Γκλόβερ και Βλαχούτιν να σχολιάσουν τις τοπικές εκλογές της Αλβανίας και κυρίως να μας ενημερώσουν για τις συστάσεις οι οποίες ε, γίνονται για να βελτιωθεί η εκλογική διαδικασία. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Γκλόβερ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε μαζί σας για τις τελευταίες ε, αλβανικές, τις δωδέκατες εκλογές όπου είχαμε παρατηρητές στην Αλβανία. Θα γνωρίζετε ίσω ότι η εκθέση δημοσιεύθηκε την προηγούμενη Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Έρχεται λοιπόν την κατάλληλη στιγμή αυτή τη συζήτηση, καθώς οι αλβανικές αρχές μας καλούν να συζητήσουμε την έκθεση και τις συστάσεις της προς το τέλος του μήνα μαζί τους. Θα γνωρίζετε ότι η FTP και η SMI έχουν δηλώσει πως είναι διτεθειμένες να τηρήσουν τις συστάσεις. Ε, σημειώνουμε επίσης ότι αυτές οι συστάσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε εκθέσεις παρακολούθησης εκλογών και στο παρελθόν χωρίς να εφαρμόσουν μέχρι τώρα. Οι εκλογές λοιπόν λαμβάνουν χώρα βάσει της νέας νομοθεσίας για τις ε, τοπικές εκλογές του 2014 για, τις, ε, για τους 61 νέους δήμους που όρισε ο νόμος για τους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους. Δημο, Ελέγχεται λοιπόν και η δυνατότητα εξαγωγή σε προσκοπτά των εκλογών αλλά και η στάση σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Βλέπουμε μια επιλογή υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο για τον ψηφοφόρο με ελευθερία έκφρασης και επιλογής, καταγραφή χωρίς προβλήματα, συμμετοχή των γυναικών και των μειονοτήτων, και τα δελικά συμπεράσματα της εκθέσεως για, για την εκλογική αναμέτρηση καταγράφουν και ε, παραθέτω ότι παρά κάποια μικροπροβλήματα το νομικό πλαίσιο θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση για δημοκρατική εκλογική αντιπαράθεση. Δυστυχώς όμως τα κύρια κόμματα ε, καταχράστηκαν των δυνατοτήτων και της θέσεώς τους κατά την εξαγωγή των, προετοιμασία και εξαγωγή των εκλογών. Συνδυαζόμενο αυτό με την πολιτικοποίηση των, ε, της εκλογικής αναμέτρησης υπονομεύτηκε ο απρόσκοπτος χαρακτήρας των εκλογών και σημαντικές πτυχέ της εκλογικής διαδικασίας θα έπρεπε να έχουν ρυθμιστεί προκαταβολικά. Δεν υπήρχε σαφήνεια ως προς την νομοθεσία και αυτό σήμανε εφαρμογή της νομοθεσίας κατά τρόπον που φάνηκε να υποστηρίζει συγκεκριμένες πολιτικές γραμμές, κομματικές γραμμές το ΣΥΣΥ, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, ε, έδρασε κατά τρόπο ανοιχτό με προγράμματα επιμόρφωσης, έλαβε ωστόσο αποφάσεις με βάση πολιτικές γραμμές και αυτό οδηγεί σε ε, παραφωνίες. Κάποιες ε, προϋποθέσεις δεν τηρήθηκαν και από τη στιγμή που η Εφορευτική Επιτροπή ήταν επικεφαλής και αρμόδια για την διεξαγωγή της εκλογικής αναμέτρησης όφιλε να προσφέρει και παρακολούθηση και επιτήρηση με κατευθυντήριες γραμμές. Έτσι δεν είχε το κοινό την εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της Φορεστικής Επιτροπής. Υπήρξε επιλογή, υπήρξε δυνατότητα επιλογής μεταξύ των υποψηφίων, αλλά η κανόνες για την καταχώρηση ενός υποψηφίου και η δυνατότητα απόστασης υποψηφιότητας ήταν τέτοιοι που δεν επέτρεπαν σε ίσους όρους κάποιος υποψήφιος να υποβάλει την υποψηφιότητά του. Επίσης τα κόμματα καταχράστηκαν και των εξουσιών και των ευθυνών τους στη διαχείριση των εκλογών, πράγμα το οποίο υπονόμευσε τις εκλογές. Υπήρξαν πολλές, ε, πολλοί ισχυρισμοί για καταχρήσεις που έφτασαν και την ημέρα των εκλογών, ισχυρισμοί για εξαγορά ψήφων για όλα, από όλα τα μεγάλα κόμματα και ως εκ τούτου για το κατά πόσο ήταν ελεύθερη ψήφος. Αξιωματούχοι από τα μεγαλύτερα κόμματα φαίνεται να αξιοποίησαν την εξουσία και τη δυνατότητες που έχουν για να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία, διανέμοντας ακόμη και ψηφοβέλτια. Ε, προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Ασάφεια και αδιαφάνεια επικράτησε ως προς την οικονομική διάσταση της εκστρατείας, όπου προβλέπεται κρατική χρηματοδότηση, ιδιωτική και δάνεια για τους ε, ε, υποψηφίους που έρχονται από κόμματα, ενώ οι ανεξάρτητοι υποψήφοι δεν έχουν δικαίωμα στην κρατική επιχορήγηση. Δεν υπήρξε λοιπόν προϋπόθεση δήλωση των δαπανών πριν από την ημέρα των εκλογών από πλευρά των υποψηφίων, ούτε και προθεσμία για την εκ των υστέρων λογοδοσία. Βλέπουμε να μην υπάρχει επαρκής παρουσία ουδέτερων και αμερόληπτων φωνών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα, ε, τους ομίλους τους, ε, του τύπου βλέπουμε μάλλον μεροληπτικές τοποθετήσεις και υποστήριξη του ενός του άλλου μεγάλου κόμματος, προβολή επίσης από τα πολιτικά κόμματα τα ίδια των πληροφοριών μέσα από τον τύπο, πράγμα το οποίο οδηγούσε σε μια ασάφεια για το ποιο, τι είδους ε, πληροφορία ήταν αυτή που κυκλοφορούσαν τα διαφήμιση, δηλαδή πολιτική ή άρθρο και σχόλιο. Η σαφήνεια δεν υπήρχε ως προστρομικό πλαίσιο και έτσι δεν υπήρξε όπως όφιλε μια διαδικασία αντιπαράθεσης στις εκλογές αυτές. Πολλές ήταν και οι προσφυγές ε, που όμως δεν ε, ικανοποιήθηκαν. Ανησυχίες υπάρχουν και για την καταμέτρηση των ψήφων που θεωρήθηκε εκρίθη εν γέννη θετικά αλλά σε μεγάλο βαθμό καταμέτρηση ολοκληρώθηκε μετά την νόμιμη προθεσμία και πολλά ήταν τα μικρά κόμματα που διαμαρτυρήθηκαν για την αδυναμία παρουσίας εκπροσώπων τους στην καταμέτρηση και εκδήλωσαν δυσπιστίες προς τελικό αποτέλεσμα της καταμέτρησης. Οι δεσμεύσει σε σχέση με τις υποχρεώσεις του ΑΣΕ και λοιπόν δεθνών οργανισμών στους οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα ε, δεν φαίνεται να έχουν τηρηθεί. Δεν υπήρχε ικανοποιητική επιλογή για τον ε, ε, ψηφοφόρο σε σχέση με την παρουσία των υποψηφίων και είναι πολύ σημαντικό για να επανέλθω στις, ε, στους του ΑΣΕ η πολιτική βούληση που εκφράζεται από τα πολιτικά κόμματα ως προς την υλοποίηση των συστάσεων του ΑΣΕ να μετατραπεί σε πράξη. Χρειάζονται και ε, κατεπηγόντως σημαντικές αλλαγές από τις συζητήσεις που έχω πραγματοποιήσει με τους κυρίους ηγέτες των, πολιτικών, των μεγάλων πολιτικών ε, κομμάτων μπορεί να γίνει αυτό. Το ODIHR δείχνει να συμφωνεί ότι θα βοηθήσει για την υλοποίηση αυτών των συστάσεων. Δηλώνει όμως ότι δεν μπορεί μόνο του να τα καταφέρει και χρειάζεται συνεργασία και άλλων κομμάτων και με τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών. Ίσως αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε στο πλαίσιο της δηλώσης ε, αρχών, διακήρυξη αρχών που είδαμε στο πίσω και την Γεωργία και το Κίεβο. Αποτελέσματα μπορούμε να περιμένουμε εάν η διεθνή κοινότητα συνεργαστεί αποτελεσματικά, συμπληρωματικά και χωρίς επικαλύψεις. Τέτοια ε, προσπάθεια λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε τώρα για να έρθουν οι κρίσιμες και κατεπίουσες αλλαγές που χρειάζεται η Αλβανία για να ε, αναπτύξει όλο το δυναμικό, πράγμα το οποίο όλοι επιθυμούμε ασφαλώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μπλάχου την έχει τώρα το λόγο και εσείς πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στις τοπικές εκλογές της Αλβανίας. Ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα βοηθήσει τις κοινέ μας προσπάθειες να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες ικανότητες στην Αλβανία για να μπορέσει στο μέλλον να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Λέδη Γλόβερ και την αποστολή της για την επαγγελματικού χαρακτήρα και πάρα πολύ αφοσιωμένη δράση τους. Μόνο μια διεθνής ε, ε, αποστολή παρατήρηση υπήρξε και προσπαθήσαμε όλοι να τη βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Συμφωνούμε απόλυτα με την ανάλυση και τι συστάσει τη έκθεση τη. Ω αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί είχαμε τον καθήκον και εξακολουθούμε να το έχουμε να τα θέσουμε όλα αυτά τα θέματα στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της ε, Αλβανίας και αν είμαστε πιο απαιτητικοί από το παρελθόν είναι γιατί έχει ανέβει ο πύχη για μια χώρα που είναι υποψήφια πριν από τις εκλογές. Κάναμε μια εξατία Συνειδητοποίησε τρία τρία κυρία θέματα. Πρώτα απ' όλα, η καταπολέμηση της οικογενειακής ψήφου που είναι κάπως ενδυμική στην Αλβανία. Ήρθαμε σε επαφή με, με αυτούς που ψηφίσουμε για πρώτη φορά, μιλήσαμε στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, παντού όπου μπορούσαμε να πλησιάσουμε τους ανθρώπους, να τους εξηγήσουμε ότι η ψήφος είναι ατομική, είναι ατομικό της δικαίωμα και πρέπει παρά τις πιέσεις που ασκούνται να την ασκήσουν ατομικά. Το δεύτερο θέμα δεν αναφέρεται σε αυτή την έκθεση, αλλά έχει να κάνει με την εφαρμογή των πολιτικών στην Αλβανία. Και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο στην Αλβανία και ελπίζουμε ότι το φθινόπωρο θα υπάρχει και ένα νομοθέτημα που θα καθορίζει καλύτερα τα του εκλέγην και εκλέγεστε ποιο έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιο και ποιο όχι. Ένα τρίτο στοιχείο που θέλαμε να κάνουμε την εκστρατεία συνειδητοποίηση είναι να οικειοποιηθούν οι πολίτε το νόημα αυτών των εκλογών. Με την παρουσία διεθνών παρατηρητών να μπορέσουν οι πολίτες να αναλάβουν ένα πιο ε, ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση και της προεκλογικής εξατίας και των εκλογών. Όλοι οι πρεσβευτέ των κρατών μελών μαζί μα ήταν ιδιαίτερα ενεργοί σε αυτό το εγχείρημα και θέλω να του ευχαριστήσω. Την ημέρα των εκλογών ήμασταν σε πολλά μέρη τη Αλβανία. Η αντιπροσωπεία πήγε σε 82 εκλογικά τμήματα. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμω είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στο μέλλον. Είναι η εφαρμογή των 22 συστάσεων και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχει μια δημόσια δήλωση πρόθεσης και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση να εφαρμοστούν αυτές, νομίζω πρέπει να αρχίσουμε αμέσως το έργο μας προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και υπάρχει μια σειρά θεμάτων τα οποία χρονίζουν, εκκρεμούν από πολύ καιρό. Είναι σημαντικό κομμάτι των πολιτικών κριτηρίων για την ένταξη της Αλβανίας και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τις βουλευτικές εκλογές του 2017. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο σαν αντιπροσωπεία κατά την απόψή μου είναι καταρχήν η αποπολιτικοποίηση της διαδικασίας αυτής. Αν διαβάσετε την έκθεση θα δείτε ότι όλα το κάθε τελευταίο στοιχείο της διαδικασίας ήταν πολιτικοποιημένο από την εκλογική επιτροπή μέχρι τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές, τους παρατηρητές κτλ. Νομίζουμε λοιπόν ότι εκεί μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει χώρος για πολίτες οι οποίοι δεν ανήκουν σε ένα πολιτικό κόμμα να συμμετάσχουν Δεύτερον, είναι η νομοθεσία για την ε, ε της πολιτικής και ένα τρίτο στοιχείο είναι το θέμα των οικονομικών θεμάτων. Το δεν έχουμε τελικά αποτελέσματα για τη χρηματοδότηση αυτών των εκλογών και τέταρτον πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη δυνατότητα στους πολίτες να παίξουν ένα πιο ένεργο ρόλο σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας και των εκλογών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Καταρχάς να δώσω το λόγο στο μόνιμο εισηγητή για την Αλβανία, τον κύριο Φλέκενστάιν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στην κυρία Γκλόβερ και στην κυρία Βλαχούτιν για την έκθεση αυτή η οποία μας δίνει μια πολύ καλή και επακριβή εικόνα για την κατάσταση στις εκλογές της Αλβανίας. Εγώ βλέπω τα πράγματα να είναι θετικά σε σχέση με αυτά που είναι πριν από δύο χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι, δεν μπορούμε, ότι μπορούμε να παραγνωρίσουμε τις παραβιάσεις που έλαβαν χώρα. Όλοι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα προβλήματα αυτά. Αναφερθήκατε σε ορισμένα θέματα, εχωρά των ψήφων, πολιτικοποίηση και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων και της χρηματοδότησης της εκστρατείας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Θα μπορούσαν ήδη να είχαν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν. Και αυτή είναι η αρνητική όψη της εκθέσεως, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα επαρκές για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, για να εφαρμοστούν συστάσεις που ήδη υπήρχαν. Και αυτό πιστεύω πρέπει να φροντίσουμε στο μέλλον το Αλβανικό Κοινοβούλιο και η Αλβανική Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το, και να επιληφθεί των θεμάτων αυτών και να εξασφαλίσει ότι οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν και εδώ περιλαμβάνεται και η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης ή από εγκληματικοποίηση της πολιτικής αν δεν μπορέσουν να επιληθούν τα προβλήματα αυτά στην Αλβανία όλες οι άλλες ε, μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να επιφέρουν, επιφέρουμε θα είναι πιο δύσκολες. Τι ερωτήματα έχω να θέσω. <clears throat> Το ένα είναι προς την κυρία Πρέσβη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της. Προφανώς θέλουμε να την βοηθήσουμε στην εργασία της. Αλλά για ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο η δικαστική μεταρρύθμιση μαζί με άλλους πρεσβευτές θα πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει ότι υπάρχει η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργήσει και να βοηθήσει. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής με αυτά που γίνονται σε επίπεδο ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο ερώτημα, απαντώντας στην έκθεσή σας μπορεί κανείς να πάρει μία από δύο ή τρεις θέσεις. Έχουμε από τη μία μεριά την κυβέρνηση που λέει εντάξει δεν ήταν πολύ καλά τα πράγματα, θα τα βελτιώσουμε. Αλλά φυσικά η κυβέρνηση θα εξάρει τη θετική πλευρά της έκθεσης. Υπάρχει αντιπολίτευση που και αυτή θέλει να διορθώσει τα πράγματα, αλλά κυρίως επικρίνει την κυβέρνηση. Το ερώτημα για μένα είναι αν τα παραδείγματα που αναφέρετε στην έκθεσή σας αν προέρχονται μόνο από τη μία πλευρά ή αν είναι ένα γενικευμένο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούκαν, ο οποίος είναι σκιώδης συγητής, έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τις δύο προσκεκλημένες μας και τις ευχαριστώ και για τις ε, αρχικές τους παρατηρήσεις και για τα όσα κάνουν ε, για την παρατήρηση των ε, αλβανικών εκλογών. Ανέκαθεν ήταν κρίσιμο το ζήτημα στην αλβανική πολιτική. Υπήρχε μία τάση οι αλβανικές εκλογές να θεωρούνται θετικές εκτός και αν υπήρχε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ στραβό. Δεν είναι σωστό αυτό. Η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα και θα πρέπει να έχουμε πολύ ψηλότερες απαιτήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, προκλήσεις για την Αλβανία, ε, αναφέρθηκαν, δεν θα τις επαναλάβω. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν όλες αυτές ε, τις προκλήσεις, υπήρχαν κάποιες θετικές πτυχές των εκλογών που ανέφερε η επικεφαλής της αποστολής παρατήρησης των εκλογών. Καταρχάς θα πρέπει να συγχαρούμε τους Αλβανούς για την υψηλή προσέλευση στις ε, ε, εκλογές ήταν 71% ε, και επίσης υπήρχε και θέμα ε, καλής εξαγωγής της προεκλογικής εκστρατείας. Όμως η τελική έκθεση των παρατηρητών καταδεικνύει ότι πρέπει να ανησυχούμε για αρκετές ελλείψεις και προβλήματα που ε, υπήρξαν σε αυτές τις εκλογές. Πάντα είναι διτό το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα στη διάρκεια των εκλογών, αλλά υπάρχουν και κάποιες πολιτικές προκλήσεις και αποφάσεις. Στην ε, έκθεση διαπιστώνω και τα δύο. Από τεχνική σκοπιά υπήρχαν αρκετά προβλήματα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για τις προθεσμίες, τις κατευθυντήρες γραμμές και την εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας, την εφαρμογή του νόμου και την ασυνέπεια των αποφάσεων ε, επίσης, ε, πράγματα που μας ανησυχούν και αυτά. Όμως ε, οι πολιτικές προκλήσεις ήταν ε, αρκετές. Ε, η πόλωση των κρατικών οργάνων που υπέσκαψαν την όλη διαδικασία, τη χρήση των πόρων για εκλογικές εκστρατείες, έλλειψη διαφάνειας, τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας και ε, έλλειψη ισορροπίας ε, στην κάλυψη των μέσων ενημέρωσης. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα και επομένως τα προβλήματα αυτά είναι πολύ σοβαρά, τα οποία ε, θα πρέπει να επιληθούν με σαφή ανάληψη πολιτικών ευθυνών. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση μου δίνουν την εντύπωση ότι οι τελευταίες εκλογές στην Αλβανία δεν μπορούν πραγματικά να θεωρηθούν ως δίκαιες και ελεύθερες εκλογές και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας επ' αυτού. Επίσης, εμένα με ανησυχεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, την ε, ποινικοποίηση των ε, πολιτικών στην Αλβανία. Ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρονολογείται εδώ και αρκετά χρόνια και ήταν και ο λόγος της τελευταίας πολιτικής κρίσης στην Αλβανία. Επίσης, ε, έρχεται να επισκιάσει και τις πρόσφατες εκλογές. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι το πρόβλημα θα πρέπει να επιληθεί μάλλον ελπίζαμε ότι θα είχε επιληθεί πριν από τις εκλογές, ε, διότι θα ήταν μια ευκαιρία για όλα τα πολιτικά κόμματα να ε, επιληθεί αυτό το ζήτημα. Παρ' όλα αυτά η ε, αντίδραση ήταν πολύ αμφίσιμη, δεν είδα καμία αντίδραση από πλευράς κυβέρνησης τους τελευταίους εννέα μήνες. Κάθε μέρα ακούμε κάποιες περιπτώσεις ε, βουλευτών με ποινικό μητρό ή ε, σκοτεινό παρελθόν που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ασυλία τους. Και αυτό φυσικά είναι ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν αρκετές συστάσεις και από τον ΟΑΣΕ και θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως οι συστάσεις αυτές. Εσείς αναφέρετε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ανέφεραν ότι σκοπεύουν να κάνουν κάτι. Ε, καλό είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πραγματικά εγώ θα ήθελα να περιμένω μέχρι να υπάρξει ε, πραγματική εφαρμογή. Καλή και η πολιτική βούληση, αλλά χρειαζόμαστε και πράξεις. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω την κυρία Γκλόβερ, Ποια είναι κατά την άποψή σας τα βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να βελτιώσουν την νομοθέτες ώστε να βελτιωθεί το εκλογικό πλαίσιο και ποια είναι τα θέματα στα οποία κατ' επανάληψη η Αλβανία δεν εφαρμόζει καλές εκλογικές πρακτικές και τα πρότυπα του ΑΣΕ. Και προς την ε, κυρία Βλαχούτιν θα ήθελα να ρωτήσω ε, το θέμα της ε, ασυλίας των βουλευτών, το αναφέρατε κι εσείς. Ε, πώς το βλέπετε εσείς από το γραφείο σας τα υπάρχει κάποια βελτίωση, μπορούμε να περιμένουμε επίλυση του ζητήματος σύντομα, ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Κούκαν, ο κύριος Φιτζίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και από πλευρά μου για την αντικειμενική εικόνα που μας παρουσιάσατε. Πολλοί ήταν οι αναλυτές που είπαν ότι οι εκλογές ε, αυτές μπορούν να δώσουν μια νέα όθηση στη πραγματεύση για ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξαν βέβαια παρατυπίες. Κυρίως ε, καταδεικνύουν την ανάγκη για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου από την Κεντρική Φορευτική Επιτροπή και πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα των πιέσεων εις βάρος των ψηφοφόρων. Για το νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν. Ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας των παρατηρητών, τι βλέπετε ως μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Κύριε Σόλτερς. Πρόεδρε. Επειδή ήμουν και μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αλβανία, στις αρχές του έτους, έξι μήνες δηλαδή πριν από τις εκλογές, μπορώ να πω ότι διαπιστώσαμε πως υπήρχαν μεγάλες και έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. είδαμε να ασκούνται πιέσει κατά τρόπο παράδεκτο, Απειλέ. Έω και βία. Έχω λοιπόν μια στιγμή ερώτηση. Η πόλωση στον πολιτικό χώρο στην Αλβανία θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες στην πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι πιστεύετε και πόσο, θα πόσο καιρό θα χρειαστεί για να βελτιωθεί η κατάσταση, πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει προκειμένου να υλοποιηθεί και η μεταρρύθμιση στο, στη δικαιοσύνη και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Τι άλλο πρέπει να γίνει μέχρι τις επόμενες εκλογές. για να γίνουν, να διεξαχθούν κατά τρόπο δημοκρατικό. Δίνω και πάλι το λόγο στις δύο προσκεκλεισμένες μας, καταρχήν στην κυρία Γκλόβερ, στη Λέδη Γκλόβερ δηλαδή. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει και τα ερωτήματά σας. Ποια είναι τα κύρια θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι τα αναφέρατε ήδη. Αλλά, όπως ελέγχεται, ένα από τα κύρια θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα αποπολιτικοποιηθούν όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στις εκλογές. Οι εκλογικές επιτροπές, τα μέσα ενημέρωσης και τα δικαστήρια. Δεν είναι κάτι το εύκολο και δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Αν υπάρχει όμως θέληση θα πρέπει να είναι δυνατόν. Και όπως είπα προηγουμένως, η διεθνής κοινότητα είναι έτοιμη να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Εξαρτάται από τις αρχές, από την κοινωνία των πολιτών και από όλα τα κόμματα στην Αλβανία να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές η, το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά, όλοι αυτοί οι φορείς θα βοηθήσουν αυτό το έργο. Δεν είναι εύκολο το έργο αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία κατ' επανάληψη έρχονται σε σχέση με τις εκλογές στην Αλβανία και αν θέλουμε λοιπόν οι εκλογές στην Αλβανία να βελτιωθούν με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε να γίνει, πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν για όλα αυτά και πρέπει να ξεκινήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Η κυρία Βλαχουτίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω τις απαντήσεις και στις τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς όσον αφορά τις ε, δυνατότητες μας ε, ως ε, διεθνούς, διεθνείς εκπρόσωποι, εμείς θα συνεργαστούμε με τον ΟΑΣΕ. Κάναμε ήδη κάποιες προκαταρκτικές ε, συναντήσεις και ε, αποφασίσαμε ήδη από το Σεπτέμβριο να προετοιμαστούμε για τις εκλογές του 2017. Δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο. Και επίσης από ότι θα υπάρξει μια ad hoc κοινοβουλευτική επιτροπή που θα ασχοληθεί με τα θέματα αυτά όσον αφορά τη δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων ε, να έχουν αποτελέσματα, νομίζω ότι εξαρτάται από την πολιτική τους βούληση. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να, κάνει, να γίνει, εξαρτάται από το αν το επιθυμούν ή όχι. Εκεί που μπορούμε σίγουρα να βοηθήσουμε είναι με την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερα ώστε να βοηθήσουμε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να εξηγήσουν στους πολίτες τι ακριβώς σημαίνει ελεύθερη ψήφος, ότι πρόκειται για ένα ε, βασικό δικαίωμα των πολιτών και όπως σας είπα έγιναν πολλές συζητήσεις και σε πανεπιστήμια και η εξαγορά ψήφων, ε, ναι μεν κάποιος ε, ε, αγοράζει μια ψήφο, αλλά κάποιος πρέπει και να την πουλήσει. Μην πουλάτε την ψήφο σας λοιπόν, διότι αυτό θα δημιουργήσει δημοκρατία στο μέλλον. πολλά λοιπόν μπορούν να γίνουν για την Αλβανία και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κατανοήσουν ποια είναι τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις τους φυσικά. Όσον αφορά τώρα την ποινικοποίηση και το να μην τιμωρούνται βουλευτέ του πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο συζητάτε αυτή τη στιγμή και οι συνάδελφοί μου επιτόπου στα Τύρανα μου λένε ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματικά καταφέραμε να θέσουμε το θέμα ε, στο δημόσιο διάλογο. Ε, ελπίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα σύντομα. Καταρχάς με τη μορφή νομοθεσίας, διότι σαφέστατα το να ε, είναι ξεκάθαρο ποιοι δεν μπορούν να είναι υποψήφοι για κάποιο δημόσιο αξίωμα και ποιοι όχι. Και αυτή είναι και απάντηση στο τρίτο ερώτημα. Ε, χρειάζεται γενικότερα μεταρρύθμιση στο τομέα της δικαιοσύνης, διότι δεν αρκούν ισχυρισμοί και απαντήσεις στους ισχυρισμούς. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που συνεχίζεται. Χρειάζεται αποτελεσματική ύπαρξη αποτελεσματικών οργάνων που θα είναι σε θέση να μπορούν να εφαρμόσουν μια ε, συγκεκριμένη νομική διαδικασία. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε κάποιους χωρίς να είμαστε βέβαιοι ότι ισχύουν ή δεν ισχύουν οι ισχυρισμοί ε, και φυσικά ε, Εκεί θα επικεντρωθούν οι προσπάθειές μας, η μεταρρύθμιση του ε, δικαστικού και του συστήματος της δικαιοσύνης και φυσικά αυτό το οποίο προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε όλους είναι ότι δεν αρκεί η νομοθεσία, ακόμα και αν είναι τέλεια, θα πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί τουλάχιστον ε, την αρχή της εφαρμογής και τη δυνατότητα της Αλβανίας να εφαρμόσει όλα όσα θα έχουν αλλάξει από πλευράς νομοθεσίας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκλόβερ έχει ζητήσει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ για να απαντήσω και κάποιες από τις άλλες ερωτήσεις. Κάποιος ρώτησε κατά πόσον μπορούμε να θεωρήσουμε ελεύθερες και δίκαιες αυτές τις εκλογές. Αυτή δεν είναι η περιγραφή που χρησιμοποιούμε εμείς ε, για τις εκλογές, ε, διότι οι εκλογές ε, είναι πολύ πιο περίπλοκες. Δεν αρκεί μια απάντηση ε, του τύπου ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Πολλές φορές ε, περιγράφεται εκλογές ως ελεύθερες αλλά όχι δίκαιες, δίκαιες αλλά όχι ελεύθερες. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε λοιπόν ε, στο εγγύς μέλλον ώστε να βελτιώσουμε τα πράγματα διότι το να συγκρίνουμε το κατά πόσον έχουν τηρηθεί κάποιες δεσμεύσεις του ΑΣΕ και γενικώ κάποιες διεθνείς δεσμεύσεις είναι αυτό το οποίο κάναμε σε αυτή την έκθεση και είπαμε ότι παρά το γεγονός ότι εφαρμόστηκαν κάποια πράγματα και υπήρξαν κάποιες αλλαγές οι οποίες είχαν συσταθεί στο παρελθόν, υπάρχουν και πολλές άλλες συστάσεις οι οποίες δεν ε, λήφθησαν υπόψη. Και αυτές είναι φυσικά αυτές οι οποίες ε, μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Ανέφερθηκα ήδη στην αποπολιτικοποίηση και συμφωνώ και φυσικά με την πρέσβυρα ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να υπάρξει μεταρρύθμιση του δικαστικού και συστήματος και της συστήματος δικαιοσύνη. Το να μπορεί κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο και να λάβει μια αμερόληπτη απάντηση ε, και να εφαρμόζεται ε, το δίκαιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεται κάποια δουλειά επ' αυτού στην Αλβανία, αλλά φυσικά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και ο ρόλος του εισαγγελέα είναι να εφαρμόζει το νόμο και φυσικά αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Ε, πολλές φορές ο εισαγγελέα εξέτασε κάποιες περιπτώσεις εκλογικών παρατυπιών, αλλά ποτέ δεν υπήρξε κάποια μερόληπτη απόφαση προς τη μία ή προ την άλλη κατεύθυνση. Και φυσικά αυτό το οποίο ε, είναι εξίσου σημαντικό είναι ο ρόλο των μέσων μαζική ενημέρωση. Οι πολίτε χρειάζονται ανεξάρτητα μέσα μαζική ενημέρωση για να μπορούν να ενημερώνονται αμερόληπτα για το τι συμβαίνει στη χώρα του. Και είναι λυπηρό το γεγονό ότι οι δημοσιογράφοι στην Αλβανία ε, λογοκρίνουν γιατί ε, είτε ε, δεν τους επιτρέπεται είτε γιατί υποστηρίζουν το τάδε πολιτικό κόμμα υπέρ κάποιου άλλου. Ε, τα πολιτικά κόμματα μπορεί να κρίνουν τις εκλογές ως καλές ή κακές, αλλά φυσικά τα πολιτικά κόμματα βλέπουν τις εκλογές από το δικό τους πρίσμα, γι' αυτό κάποιοι θα πούνε ότι ήταν καλές και κάποιοι άλλοι κακές. Αλλά όπως σας είπα ήδη, εμείς ε, με χαρά διαπιστώσαμε ότι κάποιες από τις προηγούμενες συστάσεις μας εφαρμόστηκαν, ενώ ε, μας ανησυχεί βεβαίως το γεγονός ότι κάποιες άλλες όχι και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτές ε, οι βελτιώσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα διότι το 2017 και οι εκλογές ε, δεν απέχουν πολύ επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν νέες αλλαγές στην νομοθεσία τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών ώστε οι πολίτες να μπορούν να γνωρίζουν τι προβλέπεται και πώς ε, μπορούν να εφαρμοστούν και τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι. Τώρα, πόσο καιρό θα χρειαστεί για να βελτιωθεί μια κατάσταση, ε, πόσο μακρύ μπορεί να είναι ένα νήμα. Μπορεί να χρειαστεί πάρα πολύ καιρό για να αλλάξει η πολιτική κατάσταση και η πολιτικοποίηση στην Αλβανία. Αλλά εάν όλοι ε, καλή την πίστη συνεργαστούν, τότε μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Και υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες μπορεί να γίνουν και βραχυπρόθεσμα και να βελτιώσουν στην αποπολιτικοποίηση ε, της ε, πολιτικής σκηνής στην Αλβανία. Και όπως είπα ήδη, ο ΑΣΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί άλλοι φορείς και η ίδια η κοινωνία των πολιτών θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχής να συνεισφέρουν και αυτοί μέσω της πείρας τους για να μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τις δύο προσκεκλημένες μας και για την εργασία τους επιτοπίως στον στις εκλογές και για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Αυτό είναι το τελευταίο θέμα το οποίο είχαμε σήμερα. Θα ξαναβρεθούμε αύριο στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ όλους και τους διερμηνείς ακόμα. <laughs> <laughs>